Siamo e Ας ξεκινήσουμε ακριβώς τη συνεδρίασή μας με τη συνηθισμένη προειδοποίηση. Η συνεδρίασή μας μεταδίδεται μέσω του διαδικτύου. Σημείο 1. Η οθέτηση συνταξής. στο σχέδιο που διανεμήθηκε στις 6 Δεκεμβρίου και αν δεν υπάρχουν ανστάσεις θεωρείται ότι εγκρίνεται. Στο σημείο 15 της ημερήσιας διάταξης βλέπετε την άσκηση του δικαιώματος εξέτασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο εντάχθηκε στην ημερήσια διάταξη μετά από αίτημα του συναδέλφου του κυρίου Νταφ. Μάλιστα, ο εισηγητής, ο κύριος Μάρτιν, αύριο δεν μπορεί να είναι παρόν, άρα δεν είναι δυνατόν να συζητήσουμε αυτό το θέμα, το οποίο βεβαίως είναι επίγον αλλά θα πρέπει να το αναβάλουμε για τη συνεδρίαση των μισθών το Γενάρη. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον συνάδελφο, τον αντιπρόεδρο κύριο Μαρτίνεφ, για τελεγή απόψεων για θέματα που αφορούν την ΚΟΖΑΚ. Και στο μας διάστημα θέλω να σας υπενθυμίσω ότι η Μίσσα προβλέπει μετά τη συνάντηση με τον αντιπρόεδρο, τον κύριο Μαρτίνεφ, την εξέταση δύο περαιτέρω εγγράφων. Πρώτον, το τρίτο σχέδιο έκθεσης που μας παρουσιάζει ο αγαπητότατος συνάδελφος κ. Ντάφ σχετικά με το πρωτόκολλο για την τσεχική δημοκρατία. Τρίτη εκδοχή της πρότασής του. Θα δούμε αν θα υπάρξει συνένεση σήμερα. Και δεύτερον, έχουμε το σχέδιο γνωμοδότηση Ράνσελ για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο 2017. Δυστυχώ δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διαθέσή μα, διότι σήμερα, όπω γνωρίζετε, η συνεδρίαση μα καθυστέρησε λόγω τη ε, συνάντηση με τον πρόεδρο Βαν Ρομπάι, ο οποίο μα ενημέρωσε για τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Μετά τις 6 το απόγευμα έχουμε τη συνεδρία των συντονιστών και για αυτούς ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένο. Ελπίζω πάντως να έχουμε την υπομονή και την ανοχή των διερμηνέων αν χρειαστεί να ολοκληρώσουμε τις εργασίες μας μετά τις 6.30. Δεν έχω ανακοινώσεις να κάνω από πλευρά μου, οπότε ας περάσουμε στην έκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων που ήδη έγιναν 17 και 18 Σεπτεμβρίου 2012 στις 4 Οκτωβρίου 2012 και στις 8 και 9 Οκτωβρίου του 2012 πάντοτε τα πρακτικά είναι διαθέσιμα και αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις θεωρείται ότι εγκρίνονται σύμφωνα με τη συνηθισμένη πρακτική. Βλέπω ότι ήδη έρχεται ο συνάδελφος, ο κύριος Μαρτίνεθ, είναι πάντοτε ακριβής στα ραντεβού του, οπότε να τον χαιρετήσουμε και να περάσουμε κατευθείαν στο σημείο 4. Ecco, il, il quarto punto Λοιπόν, σημείο 4 στη μισή Θα μας ενημερώσει ο Αντιπρόεδρος, ο κ. Μαρτίνεθ, για τις τελευταίες εξέλιξεις τη συνεδρίαση της ΚΟΖΑΚ. Υπάρχει παράδοση σχετικά να γίνεται αυτές οι συζητήσεις στην Επιτροπή μας και πάντοτε ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο κύριος Μαρτίν και ο παρελθόν, έχει τι μαζί μας και τον ευχαριστούμε. Τελευταία τη συνάντηση στις 19 Μαρτίου. Από τότε είχαμε δύο συνεδριάσει σε ολομελίες τη ΚΟΣΕΚ. Πρώτον στην α, Κοπενχάγη το περασμένο Απρίλιο και μια δεύτερη συνεδρίαση στην Κύπρο, στην Λευκοσία. 14 με 16 Οκτωβρίου. Και προβλέπεται μια συνεδρία των Προέδρων της ΚΟΖΑΚ για την προετοιμασία της Ολομέλειας που θα λάβει χώρα αργότερα για τις 27 και 28 Ιανουαρίου ε, στο Δουβλίνο. Επειδή η Ιρλανδία αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου το επόμενο εξάμεινο. Τα έγγραφα που αφορούν τις τελευταίες δύο συνεδριάς ολομελίας που ανέφερα ε, στην Κοπενχάγη και στην Κύπρο έχουν ήδη διανεμηθεί στα μέλη. Η συζήτηση πρέπει να είναι πολύ διότι σήμερα πραγματικά μας πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος. Βεβαίως η συζήτηση δεν χρειάζεται να περιοριστεί αποκλειστικά σε θέματα ΚΟΖΑΚ. Μπορούμε να συζητήσουμε και θέματα σχέσεων με τα εθνικά κοινοβούλια. Πάντως ο χρόνος μας είναι πολύ περιορισμένος, διότι αυτό το σημείο θα πρέπει να κλείσει το αργότερο στις 5.30. Κύριε Τιπρόεδρε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Κάρλο, αγαπητοί και αγαπητές φίλες και φίλοι. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο και την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων για την πρόσκληση αυτή. Και θα ήθελα, Κάρλο, να σου κάνω την εξή πρόταση. Θα κάνω μια σχετικά σύντομη τοποθέτηση και για διαφόρους λόγους θα ήθελα να σου δώσω την ανακοίνωσή μου, ουσιαστικά ε, με όλα τα στοιχεία, αντί να την αναφέρω προφορικά, διότι κατανοώ ότι μας πιέζει ο χρόνος. Όλοι μας, όλοι όσοι συμμετέχουμε σε όλες τις επιτροπές μας, λόγω ε, της παρουσίας του κύριου Ρομπάη, όλοι έχουμε πολύ λιγότερο χρόνο στη θέση μας. Οπότε να κάνω εδώ μια γενική τοποθέτηση, κάποια γενικά σχόλια και αύριο το πρωί να διαβιβάσω στη γραμματεία της Επιτροπής σας ε, μια πλήρη ανακοίνωση, την πλήρη αν θέλετε παρουσίαση που θα μπορούσα να κάνω με όλα τα στοιχεία που θα μπορούσα να συμπεριλάβω, στοιχεία που θα μπορούσαν ίσως να σας ενδιαφέρουν, ώστε να χρησιμοποιήσουμε τον πιο σοφό χρόνο τρόπο, συγγνώμη, το χρόνο και να κλείσουμε τη συζήτηση και νωρίτερα από το χρόνο που εσύ πρότεινες. Αν συμφωνείς λοιπόν, μια πιο πολιτική τοποθέτηση θα κάνω σχετικά με τα συμπεράσματα που μπορεί να εξάγει κανείς ε, για την τροπή που έχουν πάρει τα πράγματα το τελευταίο διάστημα και θα σας δώσω την γραπτή μου τοποθέτηση και από εκεί και πέρα, λόγω και εσείς κρίνετε τι μπορείτε να την κάνετε. Όπως είπες και εσύ, είχαμε δύο συνεδρία ολομελίας, η πρώτη τον περασμένο Απρίλιο στην ε, Κοπενχάγη και η δεύτερη στη Λευκοσία τον Οκτώβρη. Και τώρα προετοιμάζουμε την επόμενη συνεδρίαση ολομελίας που θα γίνει το πρώτο εξάμεινο στο Λούβλινο, αλλά πριν από την ολομέλεια, ήδη το Γενάρη έχουμε την συνηθισμένη προσπαρασκευαστική συνάντηση της ε, Προεδρίας, όπως λέγεται, της όλης διαδικασίας. Είναι πολύ σημαντικό να σας διαβιβάσω, αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι, το εξής μήνυμα. Τους τελευταίους μήνες δύο είναι τα γεγονότα που έλαβαν χώρα. Πρώτα απ' όλα, είχαμε μια σημαντική βελτίωση του περιβάλλοντος ε, που είχαμε στην ΚΟΖΑΚ εδώ και κάποιο διάστημα. Δηλαδή, βελτιώθηκαν οι σχέσεις Βελτιώθηκε η επικοινωνία ανάμεσα στους υπεύθυνους εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων που ε, εκπροσωπούσαν τη χώρα του ΣΤΙΚΟΖΑ και την αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, μπορεί να σημειώσει κανεί ε, ότι υπάρχει μια βελτίωση και με ικανοποιεί ιδιαίτερα αυτό το γεγονό. Και ο ίδιο ο πρόεδρο Καζίνη πιστεύω ότι μπορεί να είναι ικανοποιημένο από την εξέλιξη. Διότι αυτή η βελτίωση των σχέσεων είναι απόλυτα θετική και για τις ίδιες εργασίες μας, για την α, εκπληρώση των στόχων που προβλέπει και η ίδια η συνθήκη. Θεωρώ βεβαίως ότι αυτή η βελτίωση των σχέσεων οφείλεται σε μια πολύ συγκεκριμένη στάση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εκπροσώπων του ήταν αποτέλεσμα μια συγκεκριμένη στάση και θέση. Το δεύτερο καινούριο στοιχείο που είδαμε το τελευταίο διάστημα και που είναι σημαντικό να καταγράψουμε είναι ότι στα πλαίσια των Εθνικών Κοινοβουλίων βλέπουμε ένα όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον, αξιοσημείωτο ενδιαφέρον για να λάβουν, αναλάβουν δράση, αν θέλετε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό φαίνεται και διαρθρώνεται με διαφορετικούς τρόπους. Υπάρχουν διαφορετικές τοποθετήσεις, διαφορετικές προσεγγίσεις. Κάποιοι μέσα στα εθνικά κοινοβούλια θεωρούν ότι αυτό μπορεί να γίνει με την πολύ στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, άλλοι το θεωρούν αυτό λιγότερο ως την καλύτερη προσέξη. Πάντω, το καινούργιο στοιχείο είναι τα εθνικά κοινοβούλια εκφράζουν ένα ε, γνήσιο και όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον ότι για, την, για τα ευρωπαϊκά πράγματα και ότι πρέπει τα Ευρωπαϊκά Κοινοβούλια να συμμετάσχουν στην όλη διαδικασία για την ολοκλήρωση του Ευρωπαϊκού Οικοδομήματος. Η ΚΟΖΑΚ λοιπόν από ένα όργανο μεγάλων εντάσεων, συγκρούσεων, ρήξεων, ανάμεσα τους ευρωβουλευτές και πολλούς εκπροσώπους εθνικών κοινοβουλίων και μάλιστα και σήμερα το ζητούσα αυτό με κάποιους συναδέλφους τα εθνικά κοινοβούλια εκφράζουν όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον να συζητήσουν ευρωπαϊκά ζητήματα με τον άλλο τρόπο. Άρα λοιπόν, πρώτα απ' όλα, και στην Κοπενχάγη, αλλά κατά κύριο λόγο στη Λευκοσία, μπορέσαμε πραγματικά να διαπιστώσουμε ότι έχει βελτιωθεί αυτή η ατμόσφαιρα. Αυτό δεν το λέω απλά έτσι για να καταγραφεί στα πρακτικά συνεδρία αλλά θέλω να το κατανοήσετε και εσείς συνάδελφοι. Εγώ θεωρώ ότι αυτό οφείλεται σε μια συνειδητοποίηση και από τη δική μας πλευρά του τι πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή, μετά από μία σειρά διασκέψεων της Κόζακ, είχαμε αντιδράσει κάποιες φορές υπερβολικές αντιδράσεις. Μόλις κάποιο εθνικό κοινοβούλιο έκανε μία δήλωση εχθρική, σαφώς εχθρική προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή σαφώς εχθρική προς το Ευρωπαϊκό Οικοδόμημα, Μόλις λοιπόν είχαμε μια τέτοια δήλωση, τέτοια φύσεω, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αμέσως αντιδρούσε ζητώντας το λόγο και έμπαινε στην αντεπίθεση, αν θέλετε. Θεωρώντας πάντοτε ότι οι άλλοι κακομεταχειρίζονται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θεωρώ λοιπόν ότι εμείς ενισυνείδητα αλλάξαμε στάση. Ελπίζοντας να μην είμαστε μόνο εμείς που αλλάζουμε στάση, αλλά και οι άλλοι και τα εθνικά κοινοβούλια θα άλλαζαν στάση. Άρα λοιπόν, συνέπεια αυτές αλλαγή ήταν οι εξή. Όταν ε, ήμασταν εμείς ε, που αντιδρούσαμε έντυγε επίθεση του Εθνικού Κοινοβουλίου, τι συνέβαινε. Όλα τα εθνικά κοινοβούλια συσπυρώνονταν μεταξύ τους ε, εναντίον ημών και ακόμα και εκείνοι που είναι, είναι και ήταν πάντοτε φιλικοί προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σοπούσαν. Και οι μόνες φωνές που ακούγονταν ήταν οι φωνέ υποστήριξης έναντι εκείνων που μα μας είχαν επιτεθεί. Όταν λοιπόν αποφασίσαμε να σοπάσουμε και να μην αντιδρούμε σε οποιαδήποτε αρνητική ή εχθρική δήλωση, τελικά η συζήτηση δεν είναι μια συζήτηση ανάμεσα σε φιλοευρωπαϊστές και ε, ευρωσκεπτικιστές. Άλλαζε, αν θέλετε, η φύση της συζήτησης. Και καταφέρναμε να ακούγονται ε, πλειοψηφικά οι φωνές των φιλοευρωπαϊστών. Και βεβαίω μπορούμε να καταλήξουμε κάποια συμπεράσματα ότι συμφωνούμε με δέκα ανθρώπους και διαφωνούμε με άλλους δύο τόσο απλά. Άρα καταλήξαμε να συμπεράνουμε ότι τελικά η σύγκρουση και η αντίθεση δεν είναι ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια εν γέννη, αλλά ανάμεσα σε κάποια Εθνικά Κοινοβούλια που βλέπουν πιο ε, ευρωσκεπτική την όλη κατάσταση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όλα αυτά λοιπόν μας επέτρεψαν και στην Κοπενχάγη και στη Λευκοσία, όταν καταλή... φτάσαμε μάλλον την ψήφιση των συμπερασμάτων, οι τροπολογία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υπερψηφιστούν σχεδόν πάντοτε, κάποιε φορέ με κάποιε μικρέ τροποποίησει, αλλά πιο πολλέ φορέ χωρί καμία αντίρρηση, χωρί καμία ένσταση και θεωρώ ότι αυτό ήταν ένα πολύ ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Πλέον δεν υπάρχει η αίσθηση της απομόνωσης για το Ευρωκοινοβούλιο. Μάλλον υπάρχει αίσθηση ότι ανήκουμε στην πλειοψηφία. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό είναι πολύ θετικό από πολλές απόψεις. Από εκεί και πέρα. Είναι αλήθεια ότι τα εθνικά κοινοβούλια έχουν μια τάση κατανοητή μεν να καλούν συστηματικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι παρούσα. Εντάξει, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι παρούσα, μεν, αλλά είναι πολύ δύσκολο να κατανοήσει ακριβώς αυτό το αίτημα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εμφανίζεται ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κάθε εβδομάδα. Η Ευρωπαϊκή λοιπόν, Επιτροπή απευθύνεται προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πιστεύω λοιπόν ότι και αυτό το ζήτημα ε, επιλύθηκε σε έναν βαθμό, βελτιώθηκε και αυτό το ζήτημα, διότι η ΚΟΖΑΚ δεν είναι μόνο ένα βήμα για τα εθνικά κοινοβούλια και μόνο είναι για τα εθνικά κοινοβούλια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να, να το αναφέρουμε και αυτό και θεωρώ ότι και ο πρόεδρος ο κ. Καζίνη έχει δραματίσει ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια. Η σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με τον Επίτροπο ή του Επιτρόπου που θα συμμετάσχουν στη συνεδρία τη ΚΟΖΑ είναι πολύ σημαντικό με τι δημόσιε που θα έχουμε εκ των προτέρων ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποκτήσει μια σημαντική προβολή έναντι των Εθνικών Κοινοβουλίων, ώστε και αυτοί να εισπράξουν το μήνυμα ότι δεν μας αγνοεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αντίθετα, όπως εμφανίζεται ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τακτικά τακτικότητα, εβδομαδιαία ή καθημερινά, κάτι αντίστοιχο προσπαθεί να κάνει και ενώπιον των Εθνικών Κοινοβουλίων. Αυτό ήθελα να πω Και αυτό σίγουρα έχει εκφράσει ως ενδιαφέρον να φέρει πέρας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βεβαίως, αυτό είχε και μια άλλη συνέπεια. Σε κάθε ένα από τα σημεία της σημερινής διάταξης ήταν σημεία κλειδιά στην ΚΟΖΑΚ, πάντοτε μια διακεκριμένη προσωπικότητα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, ήταν ε, είτε ο βασικός ομιλητής, ο keynote speaker, ή τέλο πάντων είχε μια παρέμβαση. Γιατί στο παρελθόν είχαμε την παρέμβαση ενός επιτρόπου. Και τα εθνικά κοινοβούλια έκριναν σκόπιμο να είναι ο κύριος Μάρκον Χάρμπερν προκειμένου στην Κοπενχάγη, ο ίδιος ο πρόεδρος ο κύριος Καζίνη, ο οποίος έκανε μια τοποθέτηση για την, σχετικά με την έννοια της α, α, αντεστραμμένης επικουρικότητας και η κυρία Περές επίσης ήταν προσκεκλημένη στη Λευκοσία και ήταν ε, και αυτή μια βασική ομιλήτρια. Φαίνεται λοιπόν ότι μια νέα τάση η οποία πλέον α, αποτελεί πλέον πρακτική και σε κάθε λοιπόν βασικό σημείο τη ημερήσια διάταξη τη να έχουμε έναν βασικό μιλητή, έναν keynote speaker από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ώστε να εξηγεί τι συμβαίνει σχετικά με αυτό το ζήτημα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που είναι εξίσου ενδιαφέρον και επί το οποίο ε, υπήρξε πρόεδρο, αλλά θα πρέπει να υπάρξει περισσότερη πρόοδο ακόμη, είναι ότι οι πολιτικές οικογένειες, δεν μιλώ για πολιτικέ ομάδε, αλλά οι πολιτικές οικογένειες συνεδριάζουν και συντονίζονται, ίσως σε ανεπαρκή βαθμό, αλλά με κάποια τακτικότητα, ώστε να ορίσουν τις θέσεις τους. Θέλω να πω ότι οι πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συγκαλούν σε δράσεις. Φιλελεύθεροι, το Λαϊκό Κόμμα, ο καθένας. Α, το Η σαλιστική ομάδα, τέλο πάντων, όλοι μας. Στην ομάδα που ανήκουμε συγκαλούμε συνεδριάσεις όπου καλούμε και συναδέλφους από τα εθνικά μας κοινοβούλια που ανήκουν στην ίδια πολιτική οικογένεια. Θεωρώ ότι αυτό ως πρωτοβουλία θα πρέπει να γίνεται πιο συχνά και να δίδεται μεγαλύτερη σημασία σε αυτές τις προσκλήσεις. Βεβαίως, θα πρέπει να το κάνουμε μεγάλη προσοχή, ώστε να μην καλούμε πάντοτε τους δικούς μας πολιτικούς φίλους. Γιατί αυτό μπορεί να οδηγήσει σε κάποια αρνητικά συμπεράσματα και σε κάποιες αρνητικές εικόνες, θα έλεγα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, λοιπόν, να μην ξεχνάμε ότι ουσιαστικά η ΚΟΖΑΚ τα τελευταία χρόνια κρατάει μία τάση. Αυτό που ενδιαφέρονται τα μέλη της να συζητήσουν, ίσως να μην ανταποκρίνεται τα απόλυτα στον ρόλο της Κόζακ. Αυτό που ενδιαφέρει πολύ συχνά τους προσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων να συζητήσουν στην και είναι α, θέματα που είναι στην Ευρωπαϊκή Ατζέντα. Πολύ περισσότερο από άλλα ζητήματα, ζητήματα που αν θέλετε ανταποκρίνονται στο ρόλο της Κόζακ. Θέματα επικουρικότητας, θέματα επιμέρους, συγκεκριμένα, αλλά μάλλον αυτά φαίνεται δεν τους απασχολούν τόσο πολύ. Κάποιοι μπορεί να το βλέπουν αρνητικά αυτό. Εμένα προσωπικά δεν με απασχολεί, δεν το θεωρώ ότι είναι ανησυχητικό αυτό ως σημάδι. Πιστεύω ότι οι σχέσεις μας βελτιώνονται, Υπάρχει λοιπόν μια σημαντική πρόοδος στις σχέσεις μας και στις εργασίες μας που όλα γίνονται με φυσικό τρόπο. Αυτή τη στιγμή η ατμόσφαιρα στην Κώστα και είναι πολύ ειρηνική και ο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι αυτός που το αναλογεί. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει στο Δουβλίνο. Από ό,τι εγώ καταλαβαίνω, θα υπάρξει μια περαιτέρω παγί, παγίωση αυτής της τάσης. Θα ζητηθούν σίγουρα θέματα επικαιρότητα, το μέλλον της Ευρώπης, προς μια Ευρωπαϊκή Ένωση που να είναι αυθεντικά μια οικονομική νομισματική και πολιτική ένωση. Σίγουρα θα συζητηθούν τα πλέον επίκαιρα ζητήματα. Πέρα λοιπόν από τα θέματα που αφορούν αποκλειστικά και στενά την ΚΟΖΑΚ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που είναι πάρα πολύ σημαντική για όλους μας και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά γενικότερα και το Ευρωπαϊκό Οικοδόμημα, θα πρέπει να λάβει υπόψη τις εξελίξεις της δημόσιας που γίνονται αυτή τη στιγμή στα εθνικά κοινοβούλια. Θα ήταν καλό να διοργανώσει τομεακές διασκέψεις, θεματικές διασκέψεις. Πιστεύω ότι Υπάρχει αυτή η τάση και θα άρεσε, αν θέλετε, μια τέτοια κίνηση να γίνει διάσκεψη για τη γεωργία. Η δική μας λοιπόν κοινοβουλευτική ε, επιτροπή γεωργίας μας, αντίστοιχε εθνικές ε, κοινοβουλευτικές επιτροπές γεωργίας με τους αρμοδίους Ευρωπαϊκές Επιτροπής να κάνουν μια διάσκεψη. Οπότε περιοδικά, τακτικά, άλλοτε πιο συχνά, άλλοτε λιγότερο ανάλογα με το τι κρίνεται σκόπιμο. Θα ήταν καλό να έχουμε τέτοιου είδους διασκέψεις θεματικές. θέματα ασφάλεια, άμυνα και εξωτερική πολιτική είναι θέματα που ασχολούν ιδιαίτερα. Και από την άλλη είναι τα θέματα που αφορούν την οικονομική διακυβέρνηση. Αυτά είναι τα πλέον επίκαιρα ζητήματα σχετικά τώρα με το τι άλλη πληροφορία μπορώ να σας δώσω. Καταφέραμε επιτέλους να βγούμε από τα διέξοδο στο οποίο είχαμε κλειστεί χάρη στην διάσκεψη των Εθνικών Κοινοβουλίων, όπου λανσάραμε ένα νέο μηχανισμό για μία μόνιμη διάσκεψη για θέματα άμυνας, ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής. Καταλήξαμε επίσης το ότι η διάσταση ε, που έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πολύ συγκεκριμένο και πλέον υπάρχει μια σαφής διάκριση και είναι σαφής η ιδιοποιώς διαφορά ανάμεσα στο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Κοινοβουλίου, αλλά δεν είναι για τέτοια διάκριση ώστε εμεί να είμαστε οι διαφορετικοί, αλλά λειτουργούμε συμπληρωματικά. Και θεωρώ ότι είναι εξαιρετικό προηγούμενο αυτό που δημιουργείται σε μια δομή η οποία παγιοποιείται σιγά σιγά και πιστεύω ότι αυτή είναι η κατεύθυνση που έχουν πάρει τα πράγματα. Δεν θέλω να μακρηγορήσω περαιτέρω. Ιδίω σε θέματα οικονομικής διακυβέρνηση που ανέφερα πριν. Στην γραπτή μου ανακοίνωση μπορείτε να δείτε πιο ε, δομημένα και διαθρωμένα όλα αυτά τα στοιχεία. Και είναι θέματα που συνδέονται με το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο αλλά και εκεί υπάρχει πρόοδος. Και θα ήθελα κλείνοντας να αναφερθώ σε κάτι που δεν θα υπάρχει στο γραπτό μου κείμενο, αλλά θεωρώ ότι είναι θεμελιώδες και είναι καλό να το λάβετε υπόψη όσοι είσαστε εδώ παρόντες. Και να ληφθεί υπόψη και σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γιατί είναι ένα θέμα που εγώ θα το θέσω στο Προεδρείο. και στη διάσκεψη των Πρόεδρων θα το θέσω επίσης. Αντιμετωπίζουμε ένα το πρόβλημα που αφορά τις σχέσεις με τα εθνικά κοινοβούλια. Γιατί σε περισσότερες από μία περιπτώσεις βλέπουμε ότι οι συνάδελφοί μας εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά από μακρές και σκληρές συζητήσεις και αντιδικίες τελικά δεν συμμετέχουν στι συνεδριάσεις που θα έπρεπε να συμμετέχουν ή με το ρυθμό που θα έπρεπε. Στην Κόζακ καταλήγουμε εγώ και ο κύριο Καζίνη να είμαστε παρόντε. Κατανοώ ότι ο καθένα έχει βαρημένη ατζέντα και ανηλυμένε υποχρεώσει, μα όλοι μα έχουμε. Θα πρέπει λοιπόν οι πολιτικές ε, ομάδες να αποστέλουν αντιπροσωπείες αλλά τα μέλη των οποίων να συμμετέχουν πρακτικά, να είναι πραγματικά παρόντα τα μέλη σε αυτές τις συνεδριάσεις. Λοιπόν, γιατί καταλήγουμε να έχουμε συνεδριάσεις ε, πολύ ενδιαφέρουσες, θεματικές συνεδριάσεις και μα, μας συνέβη πρακτικά σε μια περίπτωση να έχουμε 40 ή 80 εκπροσώπους εθνικών κοινοβουλίων και από την άλλη πλευρά κανένας να μην εκπροσωπεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι κάτι που θα πρέπει να κατανοήσουν ε, οι πολιτικές ομάδες. Και είναι κάτι που πρέπει να διορθωθεί, να αλλάξει. Το λέω με κάθε αγάπη, σε κάθε συνάδελφο προσωπικά και στους συντρόφους της ομάδας μου. Δεν γίνεται όταν αποστέλουμε μία αντιπροσωπεία στη διάσκεψη της ΚΟΖΑΚ, μετά να απουσιάζουμε. Μα η συνεδρίαση τη ε, Κόζακ είναι σαν το Tour de France, ο κύριο τη Γαλλία. Δηλαδή είναι κάτι τόσο σημαντικό. Δεν μπορεί ξαφνικά στο τέταρτο γύρο να φύγει. Α, και να πείτε, α, ξέρετε, εμένα μου αρέσει ο, ο, ο έκτο ε, γύρο. Μπορώ. Όχι, κοιτάξτε, ή από την αρχή στο τέλο θα είσαστε ή δεν θα είσαστε. Δεν γίνεται. Κατανοώ ότι υπάρχουν και θέματα σοβαρά που μπορεί να προκύψουν ξαφνικά. Υπάρχει ανωτέρα βία, το καταλαβαίνω αυτό. Αλλά δεν γίνεται αυτή τη στιγμή ορίζεται μια αντιπροσωπεία ήδη να αρχίσουν τρει-τέσσερι και να λένε, ξέρετε, εγώ θα έρθω τη δεύτερη μέρα και θα φύγω την τρίτη μέρα. Ε, δεν γίνεται, μην πάτε τότε. Να πάει ένα άλλο που έχει χρόνο και ενδιαφέρον να κάνει αντίστοιχα και πολύ καλά την ίδια δουλειά. Πρέπει να επιτύχουμε περισσότερη πρόοδο. Και εδώ αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε πρώτα απ' όλα οι πολιτικέ ε, ομάδε. Γιατί τι κάνουμε, τσακωνόμαστε με τα εθνικά κοινοβούλια. Πολλέ φορέ. Ε, θα πρέπει τουλάχιστον οι εκπρόσωποι μα εκεί να είναι μία σημαντική εκπροσώπηση. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε εκεί και να είμαστε ένα ή δύο και σε κάποιε περιπτώσει να μην υπάρχει κανένα εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλου, θεωρώ ότι είναι σκανδαλώδε. Είναι αντιπαραγωγικό και όταν έχουμε μία συνάντηση εδώ στις Βρυξέλλες και έρχονται πάλι εκπρόσωποι των Ευρωβουλίων και πάλι δεν μας βρίσκουν. Αποσιάζουμε από την αίθουσα ή α, είμαστε για πέντε λεπτά και μετά εξαφανιζόμαστε. Δεν πιστεύω αυτή είναι η εικόνα Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ήταν κάτι πραγματικά πολύ αμήχανο και μετα ξαφανιζομαστε δεν πιστευω αυτη ειναι η εικονα ευρωπαικου αρνητικό και για μένα και τον κύριο Καζίνη να το αντιμετωπίζουμε. Γιατί ξέρετε και αυτοί που αποσιάζουν, αυτοί που τα κάνουν αυτά, φίλοι μα είναι. Αλλά το σύστημα δεν λειτουργεί. Κάτι πρέπει να γίνει και θα πρέπει αυτό να το καταγράψει και ε, η δική σας επιτροπή. Μια επιτροπή που έχει το κύρος όπως η δική σας επιτροπή μπορεί να τοποθετηθεί και να κάνει κάτι για ένα τέτοιο ζήτημα όταν έχουμε να κάνουμε δραστηριότητε που αφορούν τα εθνικά κοινοβούλια, θα πρέπει και η δική μα τάση να είναι διαφορετική και θα πρέπει η πειθαρχία και η ευθύνη να είναι κάτι που το εννοούμε. Δεν μπορούμε τώρα τέσσερα χρόνια να τσακωνόμαστε για το πού θα γίνει και αν θα γίνει η διακοινοβουλευτική διάσκεψη για θέματα ασφάλεια και άμυνα και τελικά ούτε έξι να μην πάμε. Εντάξει, άμα είναι, Α πάμε εμείς οι δυο μας πάντοτε. Εγώ θεωρώ πως το αποτέλεσμα είναι γελίο. Η εικόνα είναι γελία. Θα πρέπει να κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια. Αυτό θεωρώ, Κάρλο, ότι έπρεπε να το πω. Δεν θα το αναφέρω γραπτό στην ανακοίνωσή μου. Ήθελα απλά να το μοιραστώ σκέψη με του συναδέλφους και πιστεύω ότι είναι κάτι που πρέπει να απασχολήσει όλους τους παρόντες. για να δούμε από κοινού όλοι μαζί τι πρέπει να κάνουμε για να βελτιώσουμε αυτές τις σχέσεις, ώστε να μην αποσιάζουμε σε τέτοιες συναντήσεις όπου ζυμώνονται πολλά πράγματα και βελτιώνονται οι σχέσεις μας με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και σε κάθε περίπτωση είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις, απορίες ή οποιοδήποτε σχόλιο επιθυμείτε να κάνετε. Και τέλος να πω ότι είναι πολύ μεγάλη προσωπική ικανοποίηση να συνεργάζομαι με τον πρόεδρο της Επιτροπής σας, με τον οποίο μας διέπει ένα πνεύμα αγαστής συνεργασίας και είναι κάτι που πραγματικά μας ικανοποιεί α, ε, βαθύτατα. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ συμμερίζομαι απόλυτα όλα όσα είπατε και ιδίως ό,τι αφορά τη δική μας επικοδομητική ε, συνεργασία είναι κάτι που κάνει και πιο εύκολες τις εργασίε μας στα πλαίσια της Κόζακα. Πάντως συμμερίζομαι και, απόλυτα, και όλα τα υπόλοιπα που είπες. Θα δώσω το λόγο στου συναδέλφου που το λόγο. Δεν έχουμε όμω πολύ χρόνο, δυστυχώ. Θέλω λοιπόν να περιουσώ σε δύο πράγματα. Πρώτον, πράγματι υπάρχει ένα σημάδι ότι αυξάνει ε, το ενδιαφέρον των Εθνικών Κοινοβουλίων προς το Εθνικό Κοινοβούλιο. Να σας υπενθυμίσω ότι έλεγε το άρθρο 10 του πρώτου πρωτοκόλλου σχετικά με τις σχέσεις μας με τα Εθνικά Κοινοβούλια και επίσης αυτό που δείχνεται και στην πράξη. Καθώς αυτή η ολομέλεια συνήθως προετοιμάζεται και με την αποστολή στον ορθοποτολογείο. Απαντούν λοιπόν οι πρόσωποι των Βουλίων στις ερωτήσεις για να προετοιμάσουν και την Ολομέλεια. Στις τελευταίες συνεδριάσεις της ΚΟΖΑΚ απάντησαν όλα τα εθνικά κοινοβούλια. Όλα τα εθνικά κοινοβούλια. Και αυτό ήδη από μόνο είναι πολύ σημαντικό σημάδι. Δεν υπάρχει προηγούμενο. Και ε, κάτι άλλο που θέλω να φέρω κι εγώ και να πω ότι και πάλι συμμερίζομαι τα λεγόμενα του κύριου Μαρτίνεθ, πρέπει να βελτιώσουμε, αν θέλετε, κάποια πράγματα και σε τεχνικό επίπεδο, σε ό,τι αφορά την ε, συμμετοχή μας σε αυτές τις συνεδριάσεις, αλλά αυτό αφορά κυρίως τον συντονισμό των πολιτικών ομάδων. Είπαμε ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε πραγματικά ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα. Ε, λοιπόν, μια προσπάθεια να ξεπεράσουμε μια ένα κρατικιστικό πρίσμα από το οποίο βλέπαμε τα πράγματα, είπαμε να κάνουμε αυτή την προσπάθεια. Όμως, αυτό θα πρέπει να εμπλουτιστεί και σε επίπεδο συμμετοχή, αλλά και με μια καλύτερη προετοιμασία. Αυτές είναι οι δικέ μου σκέψεις. Θα δώσω το, λόγο στον κύριο Κουρμάη, παρακαλώ. Thank you very much, uh, President. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να θυμηθούμε ότι το 89 είχαμε ή ιδρύθηκε η ΚΟΣΑΚ και έχει επομένως κάποιο ιστορικό. Επίσης σημαντικό είναι να θυμόμαστε ότι αν δεν σεβόμαστε το παρελθόν δεν μπορούμε να έχουμε κανένα μέλλον. Αφού λοιπόν βρισκόμαστε λίγο χρόνο πριν τα Χριστούγεννα θα ήθελα να δηλώσουμε προς την Κόζακ ότι τα κατάφερε πολύ καλά, ότι πάντα μπορεί να υπάρξει βελτίωση αλλά αυτό δεν εξαρτάται από τους ίδιους. Βέβαια ζωτικό είναι ότι ο πρόεδρος μου και ο αντιπρόεδρος Μαρτίνες είπαν ότι υπάρχει πολύ καλή συνεργασία μεταξύ τους αλλά επίσης θα έπρεπε όπως επίσης είπε ο κύριος Μαρτίνες ότι και εμείς δεν ερχόμαστε εδώ απλώς για να παραστούμε αλλά για να συμβάλλουμε ενεργά γιατί συνέβη επανειλημμένος στη Βουδαπέστη να οργανώνονται εκδηλώσεις αλλά να έρχονται μόνο αυτοί οι δύο κύριοι και κανένας άλλος συνάδελφός μας. Γι' αυτό πιστεύω ότι αν δείχνουμε αυτή την εικόνα στα εθνικά κοινοβούλια τότε και εκείνα θα πάψουν να ενδιαφέρονται για μας και αυτό δεν είναι πολύ θετικό. Γι' αυτό Ευχαριστώ ιδιαίτερα για την προετοιμασία του ερωτηματολογίου που πρέπει να το εκμεταλλευτούμε δεόντως. Βέβαια υπάρχει ανάγκη μεγαλύτερη διακοινοβουλευτική συνεργασία και περισσότερο εθνικό έλεγχο και άρα η ενίσχυση του διαλόγου με την ΚΟΣΑΚ είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό αλλά αυτό το εργαλείο συνεργασίας πρέπει να χρησιμοποιηθεί πλήρως και το τονίζω αυτό το πλήρως διότι μπορεί να χρειαστεί πολύ μεγαλύτερες ε, βελτιώσεις. Και, το και τα Εθνικά Κοινοβούλια λοιπόν και το Ευρωπαϊκό πρέπει να συνεργαστούν περισσότερο, να ανταλλάξουν πρακτικές και να συζητήσουν τις αποφάσεις που λαμβάνονται εδώ μέσα. Θα ήθελα επίσης να τονίσω τα συμπεράσματα της τελευταίας συνεδρίασης του Οκτωβρίου της ΚΟΣΑΚ όπως είπε και ο Αντιπρόεδρος Μαρτίνες, για τη στρατηγική του 2020 και την έξοδο από την κρίση, συμφωνώ ότι χρειάζεται στενή εποπτεία από τα Εθνικά Κοινοβούλια για την εφαρμογή της στρατηγικής του 2020, αν θέλουμε να μπορέσουμε να αντιδράσουμε έγκαιρα και αποτελεσματικά για να βγούμε από την κρίση. Αυτός είναι ο στόχος της στρατηγικής αυτής. Εξάλλου και η κρίση δεν είναι απλώς χρηματοπιστωτική, είναι και δημοκρατική, κρίση δημοκρατίας. Είναι λοιπόν και η πολιτική διάσταση πολύ σοβαρή και πρέπει να την παίρνουμε πάντα υπόψη μας. Τα συμπεράσματα ζητούν από την Κομισιόν να ενισχύσει τη συνεργασία της με τα εθνικά κοινοβούλια γιατί χρειαζόμαστε όραμα παιδαγωγική και την κοινοτική μέθοδο. Να αυξηθεί και ο αριθμός και η ποιότητα των επαφών αυτών. Δεν ξέρω πώς ακριβώς θα μπορούσε να ενδυναμωθεί αυτός ο διάλογος, ούτε αν υπάρχει μήπως καμία έλλειψη πολιτικής θέλησης για να ενισχυθεί. Αλλά πρέπει να βρεθεί μια λύση και αφού είναι η πολύ ψηλή ποιότητα οι συνεργάτες μας, έχω ελπίδες ότι θα τα καταφέρουμε. Ευχαριστούμε κυρία Γκορμάη και τώρα ο κύριος Ντούφ. Πρόεδρε, ε, εν μέρη την αισιοδοξία του κυρίου Μαρτίνες και τον ευχαριστώ καθώς και σας για την αποφασιστικότητα και δέσμευσή σας στην υπόθεση της Κόζακ. Πρέπει όμως να καταλάβουμε όλοι ότι η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η σχέση του με εκείνη δεν είναι αυτή που θα έπρεπε. Γιατί ίσως αναπόφευκτα, διότι το ομοσπονδιακό σύστημα πολυεπίπεδων πολυεπίπεδης διακυβέρνησης που ισχύει στην Ένωση και στο Κοινοβούλιο αντικατοπτρίζεται και στις μορφές που παίρνει η κοινοβουλευτική δραστηριότητα ένα ομοσπονδιακό κοινοβούλιο μπορεί να συνεργαστεί με εθνικά για να συμφωνήσουν ορισμένα πράγματα εκ των προτέρων ή για να εποπτεύσουν την εφαρμογή των αποφάσεων από κοινού. Αλλά και αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι παραβιάζει τις δικαιοδοσίες του Κοινοβουλίου μας και των εθνικών. Δεν είναι επομένως περίεργο ότι πολλοί ευρωβουλευτές ή μάλλον εθνικοί βουλευτές εννοεί ο μιλητής ε, θεωρούν την παρουσία μας στην Κόζακ περίεργη και ανώμαλη. Θα ήταν όμως παράλογο να μην υπάρχει καμία πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ Εθνικών και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίων για αυτό το ουσιώδες θέμα. Άρα πρέπει γρήγορα σχετικά να προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε το άρθρο 13 του Δημοσιονομικού Συμβολέου ή Συνθήκης που μας επιβάλλει να βελτιώσουμε τη διακυβερνητική συνεργασία στον τομέα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Δηλαδή, να καθορίσουμε κάποια οργανωτική δομή για τις σχέσεις μεταξύ ημών και των Εθνικών Κοινοβουλίων που έχουν υπογράψει τη συνθήκη αυτή. Πρέπει λοιπόν εμείς να πάρουμε την πρωτοβουλία και γρήγορα το επόμενο έτος. Η δε συνεδρίαση του Συμβουλίου την περασμένη εβδομάδα μας ενθαρρύνει να πράξουμε κάτι τέτοιο. Ευτυχώς Το Συμβούλιο υπήρξε, εκφράστηκε ευγενός για τη δραστηριότητα των Εθνικών Κοινοβουλίων, αλλά επίσης επιβεβαίωσε την κυρίαρχη θέση που πρέπει να παίζει το δικό μας κοινοβούλιο, την πρωταρχική θέση όσον αφορά την εποπτεία των κοινών τμήματων στα δύο σώματα της διαχείρισης της χρηματοπιστωτικής πολιτικής. E Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπρόνος έχει το λόγο. Uh, Ευχαριστώ. Δεν συμφωνώ σε πολλά πράγματα με τον κύριο Μαρτίνες. Βεβαίως συμφωνώ όμως ότι αυτοί που ε, των οποίων η δουλειά είναι να και πληρώνονται γι' αυτό να πάνε σε κάποιες ε, συνεδριάσεις πρέπει να πηγαίνουν γι' αυτό συμφωνώ με αυτό που είπε πρόσφατα ο κύριος Φαρχόφστατ για τον κύριο Φάρατζ αναρωτιέμαι πώς επιλέγονται οι ευρωβουλευτές που πάνε στην Κόζακ και πώς συμφωνούν οι ευρωβουλευτές να πάνε τελικά στη ΚΟΖΕΚ. Φαντάζομαι ότι άπαξ και έχει γίνει αυτό, άσχετα αν μας ενδιαφέρει όχι το θέμα που συζητείτε, πρέπει να είμαστε παρόν, παρόντας. Αυτό ισχύει και για τις άλλες επιτροπές και για οποιοδήποτε συνεδριάσεις. Παρεπιπτόντος η ΚΟΖΑΚ είναι ένας ίσως το μόνο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο εγκρίνω όσο ζει βέβαια η Ευρωπαϊκή Ένωση η και είναι καλό πράγμα που υπάρχει. Ευχαριστώ. Πρώτα-πρώτα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Αντιπρόεδρο Μαρτίνες και τον κύριο Καζίνη για την πολύ σημαντική δουλειά που κάνουν στην Κόζα και που σίγουρα βοήθησε στο να βελτιωθεί η ατμόσφαιρα στην Κόζα και οι σχέσεις με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, ιδιαίτερα από το φως αυτών που καλούμε θα να κάνουμε ε, στο μέλλον. Μετά από την παρέμβαση του Άντριου Νταφ δεν έχω πολλά να πω γιατί και εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό το σημείο εκείνο για τη δημοκρατική λογοδοσία που περιλαμβάνεται στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ε, σίγουρα είναι γεγονός ότι η λογοδεσία και η ευθύνη ε, ε, ε, πρέπει να κρατείται στο επίπεδο το οποίο συζητεί τα θέματα αυτά και το άρθρο 13 αλλά το άρθρο 13 του Δημοσιονομικού Συμφώνου ε, ουσιαστικά δεν μας λέει ότι θα πρέπει να συζητήσουμε το θέμα της λογοδοσίας ή της ευθύνης η, αυτή, η λογοδοσία και η ευθύνη και η διαφορετική ρόλη των διαφόρων οργάνων στα διαφορετικά επίπεδα είναι δεδομένα το δημοσιονομικό σύμφωνο μας λέει να συζητήσουμε πέρα από αυτό ε, εν πάση περιπτώσει εγώ συμφωνώ με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και από αυτόν πρέπει να ε, στηριζόμαστε ε, και για τα θέματα που αφορούν την ΚΟΖΑΚ. Και μια ακόμη παρέμβαση από τον κύριο Γκουερέρο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον κύριο Μαρτίνεθ για αυτή του την διαθεσιμότητα να έρχεται τακτικά στην Επιτροπή μας και να μας παρουσιάσει και τα αποτελέσματα της ΚΟΖΑΚ Σε ό,τι αφορά μία δήλωση του κυρίου Νταφ, ήθελα να αναφερθώ. Σχετικά με την αισιοδοξία του κύριου Μαρτίνεθ, θέλω να πω, υπάρχουν πάρα πολλές έρευνες που επισημαίνουν ότι οι άνθρωποι είμαστε αισιόδοξοι στην αρχή της ζωής μας, μετά πέφτει αυτή η αισιοδοξία στη μέση ηλικία και αρχίζουμε και πάλι να είμαστε πιο αισιόδοξοι όταν αρχίζουμε να μεγαλώνουμε λιγάκι. Αυτό βεβαίω φέρτε δεν έρχεται σε σύγκρουση ε, με την κοινή λογική. Πάντως, ο Μικελάχελ είναι χρηστικό παράδειγμα ενό ανθρώπου που είναι αισιόδοξο στη ζωή και που με αισιοδοξία αντιμετωπίζει τα πάντα και στη δουλειά του. Και θέλω να το συγχαρώ γι' αυτό. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο που συνδέεται και με αυτά που είπε ο κ. Γκουαλκέρη και ο κ. Νταφ και ίσως να προσθέσω και κάτι παραπάνω. Σχετικά με τον κίνδυνο που μπορεί να υλοχεύει αυτός ο δρόμος που έχουμε πάρει εδώ στον Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, από τη μία πλευρά υπάρχει ένα πολύ θετικό κομμάτι συνεργασία με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Αυτή η συνεργασία, λοιπόν, μήπως καταλήξει να γίνει πολύ πιο περίπλοκη και δύσκολη όταν θα μπούμε στα χωράφια τη ευρωπαϊκή αρμοδιότητα, σε θέματα τέτοια που είναι ευρωπαϊκή αρμοδιότητα. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθο, αλλά αυτοί που δεν βλέπουν και τόσο θετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι α, κάποια κρατημέλη, αλλά και κυρίως είναι μέλη της δημόσιας διοίκησης. Και ίσως να αρχίσουν να προσπαθήσουν να βρουν τρόπους με τον οποίο να μπορέσει να αποδυναμωθεί ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο μέσω αυτής της συνεργασίας με εθνικά κοινοβούλια για τομεακά ζητήματα. Και με αυτόν τον τρόπο κυβερνήσει να προσπαθήσουν να υπονομεύσουν και να αποδυναμώσουν το δικό μας ρόλο. Θέλω να πω ότι κάποια στιγμή στην όλη διαδικασία Είχατε την εικόνα στο μυαλό σας ότι θα θέλατε να έχουμε τελικά ένα Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο οποίο να μπορέσουμε να αγκαλιάσουμε και μέλη εθνικών κοινοβουλίων και το αντίστροφο, ώστε κάποια ζητήματα να συζητούνται σε επίπεδο διασκέψεων στα πλαίσια μιας μικτής δομής εκπρόσωπο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Εθνικών Κοινοβουλίων. Αυτό σαν εικόνα θα πρέπει να μας κάνει να είμαστε πολύ προσεκτικοί διότι, διότι τελικά η ευθύνη, η λογοδοσία, ο δημοκρατικός έλεγχος πάντοτε γίνονται στο αντίστοιχο επίπεδο της ευθύνης του καθενός. Άρα η συνεργασία που είναι αναγκαία και πολύ καλή είναι, αλλά η επικάλυψη ανάμεσα σε θέματα που είναι ευρωπαϊκή αρμοδιότητα με θέματα που είναι εθνική αρμοδιότητα είναι κάτι που μπορεί να μα οδηγήσει σε κάτι προβληματικό και θα πρέπει να το αποφύγουμε. Ήθελα να το επισημάνω. Ευχαριστώ, Λε Λεπρόεδρο. Οπότε το λόγο τώρα έχει ο κύριο Θα Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα Σα ευχαριστώ όλου για τι τοποθετήσει σα. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για, τις, ε, για τα σχόλιά της. Και για το γεγονό ότι βλέπετε καλό να διατηρηθεί το βήμα που δίνει η Κόζα και να μπορέσουμε να τη χρησιμοποιήσουμε όσο γίνεται περισσότερο. Ο κύριος Νταφ είπε δύο πράγματα που εμένα με ασχολούν ιδιαίτερα. Πρώτον, Άντριου, δεν ξέρω κατά πόσον η ένταση μέσα στα πλαίσια μιας φιντερλιστικής δομής που βιώσαμε και εσύ ε, και εγώ, αλλά τελικά είναι πολύ μακριά ακόμη αυτό το όραμα μιας ομοσπονδιακής Ευρώπης. Δεν ξέρω λοιπόν αν είναι κάτι αναπόφευκτο ή όχι. Όταν μιλάμε για φιλοδοξίες και αρμοδιότητες των εθνικών κοινοβουλίων από τη μια πλευρά και ενός ομοσπονδιακού, αν θέλετε, κοινοβουλίου από την άλλη πλευρά. Είναι σαφές ότι θα πρέπει να ε, ορίσουμε με απόλυτη σαφήνεια τι αρμοδιότητε. Αλλά από εκεί πέρα πάντοτε θα υπάρχουν θέε ζώνε και πάντοτε θα υπάρχουν κάποιε επικαλύψει. Και όπω και πολύ ορθώ είπε και γνωρίζει και στη χώρα σου και στη δική μου χώρα, κάποιε στιγμέ, κάποιε κοινότητε θέτουν το ζήτημα των αρμοδιοτήτων και πώς διαρθρώνονται οι σχέσεις και οι αρμοδιότητες ανάμεσα σε αρμοδιότητες Ενό ε, κεντρικού κράτου με τι αρμοδιότητε που θα πρέπει να επιμεριστούν σε ένα ομοσπονδιακό κράτο. Πάντως εγώ δεν θα έλεγα ότι όλο αυτό πρέπει να οδηγήσει σε σύγκρουση και αντιμετώπιση, αλλά στα πλαίσια ενό δημοκρατικού μηχανισμού θα πρέπει να αμβλύνονται οι αντιθέσει και να μειώνονται οι αντιπαραθέσει. Επίσης είπες και εσύ και άλλοι συνάδελφοι ότι κάτι που είπε και το Ευρωπαϊκό ε, Συμβούλιο. Και έχω και τα συμπεράσματα μπροστά μου στα γαλλικά. Ένα νέο μηχανισμό που έχει σκοπό να έχει μια συνεργασία ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Εθνικά Κοινοβούλια σύμφωνα με το άρθρο 13 της συνθήκης και το πρωτοκόλλου της συνθήκης κάτι που μπορεί πρέπει να συμβάλλει σε αυτή τη δικασία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια θα ορίσουν από κοινού την οργάνωση και την προαγωγή μίας κοινή διάσκεψης του εκπροσώπους τους και να συζητήσουν τα θέματα που αφορούν την Οικονομική Νομισματική Ένωση. Αυτός δήλωση μου δημιουργεί ένα θέμα ερμηνείας. Τι σημαίνει αυτή η φράση. Σε τι αναφέρεται το Συμβούλιο. Σε μία διάσκεψη που θα συγκληθεί άπαξ και μετά ολοκληρώνει το ρόλο της ή μιλάει για μια μόνιμη δομή το Συμβούλιο όπου θα ζητήσει ουσιαστικά τα θέματα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Εγώ, εγώ θα, θεωρώ ότι λογικό είναι να εννοεί μία μόνιμη δομή, διότι αυτά τα ζητήματα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης είναι θέματα που ε, απλώνονται στον χρόνο και δεν μπορεί η συζήτηση να καλυφθεί ε, μία φορά. Χρειάζεται μία μόνιμη δομή που να παρακολουθεί σε κοινοβουλευτικό επίπεδο ή αυτό που λέτε στα αγγλικά scrutinizing να κάνει. Αυτός ο έλεγχος, ο κοινοβουλευτικός έλεγχος, που ίσως η λέξη έλεγχος να μην καλύπτει απόλυτα την έννοια του scrutinize στα αγγλικά. Πάντως είναι ότι πιο κοντά μπορούμε να πούμε. Εμείς πάντως έτσι ερμηνεύουμε αυτή τη δήλωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για μια διάσκεψη. Αυτό που ο κύριος Ρόξ, ε, να πω σας ευχαριστώ, γιατί επισημάνατε τη χρησιμότητα που έχει η κόσα και εγώ θεωρώ ότι είναι χρήσιμο όργανο σε ό,τι αφορά τους ε, εκπροσώπους μας εκεί. Να πω ότι η προσωπία στην κόσα και είναι μια αντιπροσωπεία που αποτελείται από έξι συναδέλφους. Λογικά οι δύο μεγάλες ε, ε, ομάδες παίρνουν τις τρεις αυτές και μετά οι υπόλοιπε ομάδες εκ περιτροπής μπορούν να αποστέλουν εκπροσώπους. Οπότε δεν εκπροσωπούνται πάντοτε όλες οι πολιτικές ομάδες. Αυτό που ο κ. Κουαλτιέρη τώρα. Συμφωνώ μαζί σας. Και εγώ θεωρώ ότι κίνουμε στη σωστή κατεύθυνση. Αυτή η σωστή κατεύθυνση όμως απαιτεί και το εξής το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παρακολουθεί στενά και καθημερινά τα πράγματα και να είναι παρόν. Γιατί είναι και θέμα εικόνα αν θέλετε. Είναι θέμα τη εικόνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, έναντι των Εθνικών Κοινοβουλίων. Και σε σχέση με αυτά που είπε ο κύριος Γκερέρο, για αυτό τον κύκλο που κάνει στη ζωή η αισιοδοξία, θεωρώ ότι είναι καλό πράγμα να είναι κανεί και χαίρομαι ιδιαίτερα ε, που επιβεβαιώνω και παληθεύω αυτή τη θεωρία που αναφέρατε. Από κάποια λίγη και μετά μας είπατε θα είμαστε όλο και πιο αισιόδοξοι. Ε, χαίρομαι λοιπόν αν μπορεί αυτό να επαληθευτεί. Πάντως, Ενρίκε, τώρα επί της ουσίας, να πω το εξή. Εμένα δεν με απασχολεί να υπάρξει ε, εμβάθυνση της τομιακής συνεργασίας. Δεν είναι κακό αυτό. Αρκεί να μην αρχίσουν να υπάρχουν προκλήσεις. Να αντικαταστήσουμε, όπως είπες και εσύ, να αντικατασταθούν οι ευθύνες και οι αρμοδιότητες. Οι ευθύνες και οι αρμοδιότητες είναι σαφώς επιμερισμένες. Και αυτό θα πρέπει να είναι σαφώς δηλωμένο και, ε, αν θέλετε, είναι κάτι παγιωμένο, δεν, δεν μπορεί να αλλάξει για παράδειγμα. Μιλάμε όμως για θέματα γεωργίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα Εθνικά Κοινοβούλια δεν μπορούν κάποια χρονική στιγμή να κάνουν μια συζήτηση, μια κοινή, πολύ ισχυρή συζήτηση για την κοινή αγροτική πολιτική και τη συζήτηση που γίνεται σήμερα για την ΚΑΠ. Αυτό δεν μπορούσε ποτέ να είναι αρνητικό, να θεωρηθεί κάτι αρνητικό. Και αυτοί που παρακολουθούν στατιστικές συζητήσει στα Εθνικά Κοινοβούλια δεν έχουν κάτι να χάσουν να συνέλθουν σε μια κοινή συνεδρίαση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπάρχει ένα θέμα ε, κοινή αντίληψη, πιστεύω, σε κάποια ζητήματα και ε, κοινή λογική. Και ένα τελευταίο σχόλιο. Και συνδέεται με αυτά που είπε ο κ. Μπρόγκ. Να μην μπερδευόμαστε. Υπάρχει ένα πρόβλημα σε κάποια εθνικά κοινοβούλια, όπου υπάρχουν πολύ ισχυρέ δυνάμει που ριζικά είναι αναφαρδόν κατά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό είναι δεδομένο, είναι μια συγκεκριμένη θέση. Θεωρούν ότι θα πρέπει ουσιαστικά να εξαλειφθεί από προσώπου γη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, εκεί έχεις ε, έναν τείχο μπροστά σου. Οπότε λογικά υπάρχει μια αντιπαράθεση. Δεν μπορείς να ξεπεράσει Είναι ένα διέξοδο αυτό ανάμεσα όλους εμάς που είμαστε υπέρ της ολοδικασίας υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις. Μπορεί να καταλήξουμε και σε επιμέρους ζητήματα να διαφωνούμε απόλυτα. Αλλά εκεί που δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συνεννόηση, ανάμεσα σε αυτού που πάνε σε συνάντηση εξ ονόματο Εθνικών Κοινοβουλίων για να δηλώσουν πολύ απλά ότι αυτό που θέλουν και επιθυμούν είναι να εξαφανιστεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Φανταστείτε, αν λέγαμε κι εμεί το αντίστοιχο, που δεν το έχουμε πει ποτέ βεβαίω. Και να πω κάτι ακόμη, Ενρίκε. Αλλά δεν θέλω να καταγραφεί στα πρακτικά. Το πρόβλημα που υπάρχει με την Κόζα και τα εθνικά κοινοβούλια, αν γένεια, είναι ότι όχι ότι υπάρχουν εθνικά κοινοβούλια ή πολύ σημαντικέ πολιτικέ ομάδε που είναι κατά της, ε, του ευρωπαϊκού οικοδομήματο. Το πρόβλημα που είναι ότι κάποια εθνικά κοινοβούλια και μέσα σε αυτά κάποιες φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις στα λόγια, τελικά στην πράξη επιδεικνύουν μια πολύ επιθετική στάση έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και υπάρχει μια ανακολουθία ανάμεσα στα λόγια και στις πράξεις. Και θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να βγούμε από αυτό το φαύλο κύκλο των πολιτικών οικογενειών. Ε, που είπατε και Εσύ φίλε μου που είσαι από την ίδια πολιτική οικογένεια, από την ίδια τη χώρα με μένα, έρχεσαι εδώ στο κοινοβούλιο και μας επιτίθεσαι. Δεν γίνεται αυτό. Είναι αδιανόητο αντίκειται ε, και σε ό,τι πιστεύει η ίδια η χώρα σου, αλλά και η ίδια η πολιτική σου ε, οικογένεια παράδειγμα κάποιες βρετανικές ε, ε, τάσει και δυνάμει που υπάρχουν και στους κόλπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλου. Μα αυτό είναι θεμητό, είναι λογικό, είναι η θέση του καθενό. Το πρόβλημα κυρίω προέρχεται από κάποιε φιλοευρωπαϊκέ πολιτικέ δυνάμει που κατά κάποιο παράδοξο τρόπο επιδεικνύουν μια τεράστια επιθετικότητα ενάντια ε, στο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλου. Αυτή είναι μια πραγματικότητα που πρέπει να καταγράψουμε. Είναι μια πραγματικότητα που ζούμε και προσπαθούμε να την αντιμετωπίσουμε. Μέσω, όπως είπα, α, αυτής ε, της νέας δομής που θέλουμε να δημιουργήσουμε μέσω των πολιτικών οικογενειών. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας ε, και για την υπομονή σας και για την πρόσκλησή σας σε κάθε περίπτωση. Και ελπίζω να συνεχίσουμε να έχουμε τέτοιου είδου ε, συναντήσει. Βεβαίω, ευχαριστώ. Εγώ σε ευχαριστώ για τη συμμετοχή σου και για τι παρατηρήσει σου, που ήταν απόλυτα πλήρε, όπω και για το γραπτό κείμενο που θα μα στείλει για να το διανύμουμε σε όλους τους ε, συναδέλφους. Αυτά και να σε αποχαιρετήσουμε. Περνάμε στο σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης. Σχέδιο πρωτοκόλλου για την εφαρμογή του χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τσεχική Δημοκρατία. Γνωρίζετε ότι ο κύριος Νταφ έχει αναλάβει αυτό το ρόλο που στην ε, μη, πρώτη ψηφοφορία δεν κατάφερε να ψηφιστεί. Στη δεύτερη ε, προσπάθειά του είχαμε μία ισοψηφία υπερκεκάτα και τώρα ελπίζουμε σε αυτό το τρίτο σχέδιο που θα παρουσιάσει να μπορέσουμε να βρούμε ένα, α, μία λύση, ένα διαξόδο. Λοιπόν, λίγο είναι ο χρόνο που απομένει, γιατί θα πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα στην ένταση των μισθών. Παρακαλώ, τον λόγο έχει ο κύριο Νταφ. Yes, uh, as you, uh... Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Όπως είπατε, αυτή είναι η τρίτη απόπειρα να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα εδώ στην Επιτροπή τα οποία θα μπορέσουμε να προωθήσουμε στην Ολομέλεια για το θέμα αυτό του τσεχικού πρωτοκόλλου που έχει συμφωνηθεί από πολιτικά από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ζητείται όμως επισήμως και γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ε, η συνθήκη και η νομολογία μας υποχρεώνει να κάνουμε αυτή τη γνωμοδότηση, να πάρουμε θέση. Για εκείνους που για πρώτη φορά συζητούν το θέμα, να πω ότι το πρώτο πρωτόκολλο αυτό είναι το πρωτόκολλο 30 της συνθήκης όπου η τσεχική δημοκρατία θα ε, πάρει την ίδια θέση με το Ηνωμένο Βασίλειο και την Πολωνία σχετικά με τον σεβασμό των ανθρωπίνων του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ε, το θέμα είναι ευαίσθητο και λεπτό. Γι' αυτό άλλωστε η Επιτροπή μέχρι τώρα δεν μπόρεσε να καταλήξει σε συμπεράσματα. Θα ήθελα απλώς να αναφέρω τις αλλαγές που έκανα στην τρίτη αυτή έκθεση σε σχέση με τη δεύτερη έκθεση. Δεν πιστεύω ότι τώρα εδώ θα πρέπει να μπούμε σε μεγάλη συζήτηση για τα υπέρ και τα κατά του πρωτοκόλλου. Να πω ότι στο προνήμιο, στο σημείο και ε, έκανα κάποια αλλαγή, έλαβα υπόψη τη θέση των πρασίνων στο παρελθόν που είχαν πει παλιότερα ότι είναι πολύ σημαντικό να καταλήξουμε σε συνένεση για το θέμα της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε όλα τα κράτη-μέλη. Έβαλα λοιπόν εδώ δύο επιπλέον λέξεις για να μιλούμε για ίση, ισότιμη εφαρμογή και εδώ ο κύριος Χέφνερ ε, θα υποβάλει φαντάζομαι κάποια τροπολογία. Τώρα, παρακάτω, στο S, άλλη αιτιολογική σκέψη, προσ, πρόσθεσα κάτι το οποίο επανειλημμένα έχουμε συζητήσει αλλά ποτέ δεν είχε εκφραστεί γραπτά. Το Ποιο δηλαδή, το ότι θα ήταν μη σόφρον για τα άλλα κράτη-μέλη να ξεκινήσουν μια να ξεκινήσουν την μεγάλη και επίπονη διαδικασία αυτή της κύρωσης του τσεχικού πρωτοκόλου πριν να είναι σίγουρο ότι η ίδια η τσεχική δημοκρατία συμφωνεί και θα προχωρήσει σε κύρωση. Συμφωνώ λοιπόν με αυτό ότι άλλες χώρες δεν πρέπει να προτρέξουν και γι' αυτό βάζω εδώ, προσθέτω εδώ ορισμένα πράγματα ότι πρώτα πρέπει να είμαστε σίγουροι για το ότι υπάρχει σαφής πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο της Τσεχικής Δημοκρατίας για την κύρωση του πρωτοκόλου αυτού πριν να αρχίσουμε εμείς να ξεκινήσουμε τις διαδικασίες ε, στις χώρες μας. Ο πρόεδρος Κλάς, Κλάς θα αποχωρήσει από τη θέση του πολύ σύντομα από τη θέση του Προέδρου δεν, πιστεύω ότι θα εξαφανιστεί από την πολιτική ζωή στην Τσεχική Δημοκρατία βεβαίως αλλά δεν θα έχει πλέον τη θέση που έχει αυτή τη στιγμή και η αποχώρηση του μπορεί να επηρεάσει την απόφαση που θα πάρει το Τσεχικό Κοινοβούλιο. Επίσης, διάγραψα ένα μια αιτιολογική σκέψη που είχαμε στο παρελθόν σχετικά με την κροατική προσχώρηση, με την ένταξη Κροατίας. Πιστεύω ότι δεν χρειάζεται, γιατί δεν νομίζω ότι χρειάζεται να συνδέσουμε ε, κάποια ε, συνδέσουμε το θέμα αυτό με ενδεχόμενη αποτυχία μας να εγκρίνουμε το, ορισμένα πράγματα σχετικά με την ένταξη της Κροατίας. Επίσης, παρακάτω προσέθεσα κάτι που λέει ότι Ε, θα πρέπει να προσέξουμε πολύ πριν γνωμοδοτήσουμε έστω και θετικά προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Εκείνο που είναι σημαντικό είναι ότι έγινε η διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην τελευταία παράγραφο, στη δεύτερη παράγραφο, αποσαφηνίζω ότι το ψήφισμα αυτό ουσιαστικά είναι η γνωμοδότησή μας ε, και παρουσιάζει τη θέση μας όπως απαιτεί η συνθήκη. Πρέπει βεβαίως να ορίσουμε και μια ημερομηνία για την κατάθεση των ε, τροπολογιών. Ελπίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Ε, ελπίζω οι συνάδελφοι να δείξουν υπομονή και ανοχή ε, στο το γεγονός ότι για τρίτη φορά που πειρώμαι να περάσω το θέμα αυτό ε, εστέ γενναιόδοροι, είμαι σίγουρη ότι είστε, είναι και Χριστούγεννα. Ε, Ευχαριστώ κύριε Τώρα δυστυχώς είμαι υποχρεωμένο να σας πιέσω χρονικά γιατί έχω πέντε αγορητές και πρέπει να απαντήσετε. Ε, και πρέπει να συνεδριάσουν οι συντονιστέ και υπάρχει και ένα άλλο σημείο. Σα παρακαλώ λοιπόν να είσαστε πολύ σωστικοί. δύο λεπτά το πολύ ο καθένα. Ο κύριο Πρατάν. Pane předsedo, děkuji za slovo. Nejprve bych chtěla poděkovat Ευχαριστώ. Το ευχαριστήσω τον εισηγητή για την όλη προσπάθεια που κατέβαλε και για την στέξη αυτό το κείμενο. Θέλω να πω ότι εντάχει ότι η θέση της γερουσίας της Δικής Δημοκρατίας παραμένει ίδια. μετά τον Οκτώβρη αυξάνει ο αριθμός των σωστελμικωτών γερουσιαστών μας που υποστηρίζουν την προσχώρηση σε αυτή τη συνθήκη. Οπότε Θέλω να αναφερθώ και στην παράγραφο που μιλάει για την ε, προτέρα προσχώρηση ε, και την επικύρωση της ε, συνθήκης από την Λοιπόν, υπάρχουν κάποια υπεροσημεία που μπορούμε να δούμε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιστεύω ότι θα πρέπει να ξαναδεί την κατάσταση και όσα έγιναν την τελευταία τριετία στη χώρα μας και να μην συζητήσει αυτόν τον αποκλεισμό λόγω των ίσων δικαιωμάτων που θα πρέπει να φέρουν όλου του πολίτες. πολίτε. Ευχαριστώ πολύ και γιατί ήσασταν πολύ σύντομοι. Η κυρία Σερκόβα. Děkuji, pane předsedo. Já budu mít trochu odlišný názor než moje předřečnice. Eh, Η θέση μου διαφέρει σε έναν βαθμό σε σχέση με την προλαλή σας. Η τρίτη εκδοχή αυτή τη έκθεσης είναι πολύ πιο θετική, κατά τη γνώμη μου πάντοτε. Αυτή είναι η θέση του ε, Δημοκρατικού κόμματο τη χώρας και θέλω να κάνω και κάποια επιμέρους σχόλια ε, για το προήμιο. Σε κάποια σημεία αναφέρεται ο κύριο Νταφ, στο Τζέι για παράδειγμα, το οποίο λέει ρητά ότι η μόνη συνέπεια του πρωτοκόλλου παριθμών 30 είναι η έλλειψη ασφάλειας δικαίου, όχι μόνο στη Τσεχία, αλλά και σε οποιοδήποτε κράτο τη Ένωση. Νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι από αυτού. Είμαστε όλοι νομικοί και δεν μπορώ να πιστέψω ότι το Κοινοβούλιο μπορεί να δεχθεί μια τέτοια δήλωση. Έπειτα στο ΚΑΠΑ λέει το πρωτόκολλο παριθμών 30 γύρει ανασφάλεια δικαίου και πολιτική σύγχυση. Ελπίζω τουλάχιστον οι δηλώσει μου να μεταφραστούν ορθά στα αγγλικά από τα τσεχικά. Δεν πιστεύω ότι μπορούμε να μιλούμε για ασφάλεια δικαίου και για πολιτική σύγχυση από προκύπτει αυτό από το γεγονός ότι η Επιτροπή μας συζητά την τρίτη εκδοχή της ίδιας έκθεσης που αφορά μόνο τη συνταγματική τάξη στην τσεχική δημοκρατία. Ω νομικός, γνωρίζοντας και τον χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων, θεωρώ ότι η θετική εκδοχή είναι πολύ πιο ακριβής και το συνταγματικό μας δικαστήριο ακριβό χρησιμοποιεί αυτή την ακριβή εκδοχή. Η μόνη λοιπόν περίπτωση σύγχυση είναι η εξή. Τελικά αυτό το πρωτόκολλο θα υιοθετηθεί ή όχι. Αυτό είναι αν θέλετε και κάτι που με παρηγορεί σε αυτή την περίπτωση. Το δεύτερο που θέλω να, να πω είναι στην παράγραφο S. Θα σπρώνω να είστε πιο σύντομοι, λέει ο πρόεδρος. Ναι, ναι, ένα τελευταίο σχόλιο. Πρόεδρε, το συγγνώμη. σχετικά με τη βούληση του Τσεχικού ε, ε, Κοινοβουλίου. Αυτή η αναφορά. Θεωρώ ότι ούτε η Επιτροπή μας, ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εν γέννη μπορεί να προκαταλάβει τη θέση του Σεχικού Κοινοβουλίου. Δεν πρέπει να παίζουμε με νομικές παραδοχές εδώ. Δεν είναι σωστός τρόπος προσέγγισης. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και ευχαριστούμε τον εισηγητή και τον πρόεδρο που μου έδωσε πλέον χρόνο. Ευχαριστώ. Κύριος Μπρόνς. Uh, Κοιτάξτε, φαίνεται από την απόφαση του δικαστηρίου πριν από ένα χρόνο καθαρά ότι το πρωτόκολλο 30 δεν χορηγεί εξαίρεση στο Ηνωμένο Βασίλειο όπως ισχυριζόταν ο Τόνι Μπλερ Το δικαστήριο είπε ότι στόχος του πρωτοκόλου 30 ήταν να εξηγήσει το άρθρο 51, αλλά δεν είναι φαρφανές γιατί το Ηνωμένο Βασίλειο και η Πολωνία χρειάζονται τέτοια εξήγηση και οι άλλοι όχι. Ίσως γιατί είναι πιο ανόητοι. Πριν από δύο μήνες δηλώθηκε ότι η χάρτα δεν χορηγεί περισσότερες δικαιοδοσίες εθνικές από την Πολωνία και τον Ηνωμένο Βασίλειο στην Ένωση. Αλλά αυτό μπορεί να, πρέπει να ισχύει και για άλλες χώρες μέλη. Πρόκειται στην ουσία όντως για μεταφορά εξουσίας από τις χώρες στην Κομισιόν. Προσπάθησε λοιπόν ο εισηγητής να ξεκαθαρίσει τα πράγματα και αν δεν το κατάφερε δεν φταίει ο ίδιος. Είναι η φύση του αντικειμένου που είναι ασαφής. Το πρωτόκολλο και εδώ διαβάζω αυτά που είπε ο κύριος Νταφ, έχει νόημα μόνο αν η χάρτα προσθεθεί στην υπάρχουσα νομολογία για να μειώ... σε περίπτωση μείωσης ε, φανερής των δικαιωμάτων, των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αλλά βέβαια θα ήταν παράλογο να μην υπήρχε κάτι τέτοιο, δηλαδή μην προστίθεται στην εθνική νομοθεσία. Δηλαδή είτε δεν έχει νόημα ε, αν αποτύχει είτε εάν πετύχει όπως λέει ο κύριος Νταφ πρέπει να χορηγεί εξαιρέσεις. Φαίνεται ότι το πρωτόκολλο θα αρχίσει να ισχύει όταν θα προσθεθεί επίσημα στο αγγλικό δίκαιο η χάρτα και ε, δεν θα είναι μία απλή μεταφορά όπως γίνεται για τις άλλες οδηγίες κλπ. Ο στόχος της ποιος ήταν λοιπόν η παραπλάνηση των μελών του Ευρωπαϊκού και Πολωνικού Κοινοβουλίου. Είχαμε συμφωνήσει σε μια διακυβερνητική διάσκεψη που δέχτηκε τη συνθήκη της Λισαβόνας και της οποίας υπάρχουν πρακτικά. Θα ήθελα να ρωτήσω από τα πρακτικά ποιος πρότεινε αυτό το πρωτόκολλο είτε ο Τόνι Μπλερ άθελά του ή θελημένα παραπλάνησε το Βρετανικό Κοινοβούλιο είτε κάποιος παραπλάνησε τον Τόνι Μπλερ. Δεν να τελειώνετε παρακαλώ. Ναι, με συγχωρείτε που με Τελευταίος, σύντομα και εκείνος, ο κ. Σέπφλινγκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι όντως σύντομος. Ο κύριος Ντάφο, όπως πάντα, μας περιέγραψε τα πράγματα με μεγάλη σαφήνεια. Μπορούμε να πούμε νομίζω ότι η πολιτική κατάσταση στην Τσεχία είναι λιγότερο ρευστή τώρα από ό,τι προηγουμένως. Η τωρινή κυβέρνηση φαίνεται ότι θα παραμείνει, θα εξαντλήσει την εντολή της και οι επόμενες εκλογές θα αλλάξουν την ατμόσφαιρα που κυριαρχεί περί του πρωτοκόλου. Το πιο σημαντικό ήταν η πρότασή σου, Ανδρέα, ότι φρόνιμο θα ήταν οι χώρες μέλη να μην κάνουν την επικύρωσή του μέχρι να συμπληρωθεί η τσεχική διαδικασία. Η διατύπωση δε ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι έχουμε τύχη διαβούλευσης μου φαίνεται σωστή. Πόσο το εξετάζουμε κανένα χρόνο ε, μάλλον θα καταλήξουμε τελικά σε κάποια συμφωνία. Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο τον νέο Ο κύριος Ντούφ, αλλά και εκείνο σύντομα. Ευχαριστώ όσους σχολίασαν. Η κυρία Τσεσκόβα έθεσε ερωτήματα που έχουν απαντηθεί αποτελεσματικά από τον κύριο Μπρόνς. Δηλαδή, το πρωτόκολλο αυτό δημιούργησε πολιτικές αναταραχές από την αρχή και είναι περίεργο ότι οι Βρετανοί και οι Πολωνοί το είδαν από αντίθετες απόψεις και θέσεις. Οι Βρετανοί ανησυχούσαν γιατί ήθελαν να μειωθεί η χρήση της χάρτας στα Βρετανικά δικαστήρια. Η Πολωνία όμως ήθελαν να επιβεβαιωθεί η σημασία της χάρτας. Το αντίθετο δηλαδή ο κεντρικός χαρακτήρας της. Μίλησα με το τσεχικό συνταγματικό δικαστήριο στο Πρνό και νομίζω ότι είδα, ήδη είδα αμφιβολίες ως προς το νόημα του πρωτοκόλου, μεγαλύτερες από ό,τι διαπίστωσα από τον κύριο Σφάρτσενπεργκ που τον εκτιμώ ιδιαιτέρως ή από την κυρία Τσεσκόβα. Θα δούμε λοιπόν, θα δούμε. Αν μπορέσουμε να καθορίσουμε, μπορούμε να καθορίσουμε κύριε Πρόεδρε προθεσμία τέλη Ιανουαρίου ας πούμε. Για τις τροπολογίες 8 Ιανουαρίου, όχι 17 Ιανουαρίου, ε, 12η Μεσημβρινή. Και επειδή ψηφοφορία μπορεί να γίνει στις 19 ε, Φεβρουαρίου στην τακτική μας συνεδρίαση. Ωραία, καλώς. Σας ευχαριστώ όλους για το λόγο. Οπότε γρήγορα πάμε στο τελευταίο σημείο της διαταξής. Στο σημείο 6, Ευρωπαϊκό Εξάμερο του Συντονισμό των Οικονομικών Πολιτικών. Γνωρίζουμε ότι εν προκειμένου αρμοδιότητα κατά κύριο λόγο έχει η Επιτροπή ΕΚΟΝ, προκειμένου εκπονούμε γνωμοδότηση, ο συνάδελφο ο κύριος Σανζέλ έκανε σκόπιμο να συμβάλλει με μια γνωμοδότηση για αυτό το θέμα. Να δώσουμε κατευθείαν το λόγο στον συνάδελφο. Πρέγω. Chairman, Κύριε Πρόεδρε, αλλά σε εξέλιξη θα φύγουν οι διερμηνείς. Ναι. I'm being assured that they're here till 7, is that correct? Μέχρι τις 7 μου λένε ότι πράγματι. Sì, come, sì, come, come ho detto all'apertura del... Όπως είπα κατά την έναρξη των εργασιών μας, ήδη εξέφρασαν τη διαθεσιμότητά τους στις 7 το απόγευμα. Οι διερμηνείς τους ευχαρίστηκαν των προτέρων, τους ευχαριστώ και πάλι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε γρήγοροι σε κάθε περίπτωση. Κύριε Ρανσέλ, έχετε το λόγο. Παρακαλώ, ενημερώστε μας σχετικά. Παρουσιάστε μας το σχέδιο γνωμοδότηση. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Πρόεδρε, κύριε Καζίνη. Θα είμαι πρακτικός στην προσέγγιση μου, γιατί αυτή η γνωμοδότηση για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο ουσιαστικά άπτεται πολλών θεμάτων τα οποία έχουμε συζητήσει και ζητούμε συνεχώ και τα οποία δεν έχουμε επιτύχει στον επαρκή βαθμό που θα θέλαμε. Ουσιαστικά η γνωμοδότηση ασχολείται με σταγματικά στιγμή. δηλαδή δεν μπαίνουμε επί της σε οικονομικά ζητήματα, ούτε μπαίνουμε σε ανάλυση των προτεραιτήτων της δημοσιονομικής και οικονομικής ε, πολιτικής, διότι αυτά είναι θέματα αρμοδιότητας Επιτροπής ΕΚΟΝ. Εμείς εδώ φύγουμε καθαρά και μόνο σταγματικά ζητήματα, θεσμικά ζητήματα, που απορρέουν από αυτό το ζήτημα θα ήθελα λοιπόν να επισημάνω εν προκειμένου σε αυτό το πλαίσιο τρία-τέσσερα σημαντικά ζητήματα. Πρώτον, είναι πολύ σημαντική η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, περισσότερη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πιο συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά τον έλεγχο της προετοιμασίας και παρακολούθηση, ένα monitoring της, της έκθεσης ανάπτυξης και στις συγκεκριμένες συστάσεις που απευθύνονται στα κρατημένη. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό, κατά πρώτο λόγο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμμετέχει στον καθορισμό των προτεραιοτήτων και πολιτικών στόχων. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχει προτέρα διαβούλευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν δημοσιεύεται η αιτήσια αυτή η έκθεση, να μπορεί επίσης να γίνει ψηφοφορία στην Ολομέλεια αυτού του εγγράφου, ώστε να σαφίσει η θέση ε, του Κοινοβουλίου προκειμένου και τέλος ή δυνατόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υιοθετεί στην αρχή κάθε θητείας του ένα έγγραφο που να ορίζει τις πολιτικές πρωτεβουλίες για την επόμενη πενταετία. Άλλο σημαντικό θέμα το οποίο ήδη ε, περιλαμβανόταν και στην περσινή γνωμοδότηση αφορά τον, ε, τον ρόλο των Εθνικών Κοινοβουλίων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει ένα διακοινοβουλευτικό διάλογο, προκειμένου, άρα θα πρέπει να υπάρχει μια σχέση ανάμεσα στα Εθνικά Κοινοβούλια με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτό το ζήτημα και πάρα πάρα πολύ σημαντικό σημείο και επέμενα πάντοτε ευθύ εξ αρχής, γιατί είναι μείζονο σημασίας είναι ότι μαζί με τα κράτη-μέλη να ασκήσουμε ένα παιδαγωγικό ρόλο, ώστε τα κοινοβούλια να υιοθετούν εσωτερικές διαδικασίες τέτοιες, ώστε να τους επιτρέπει να συμμετέχουν ενεργά κατά την κατάρτιση των εθνικών μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων σε καμία περίπτωση δεν προτείνουμε τον περιορισμό των αρμοδιοτήτων των Εθνικών Κοινοβουλίων. Ζητούμε αλλαγή των χρονοδιαγραμμάτων των Εθνικών Κοινοβουλίων. Θα πρέπει δηλαδή νωρίτερα να παρεμβαίνουν στη διαδικασία για την προετοιμασία του εθνικού προλογισμού και να κάνω μια συζήτηση σε δύο χρόνους. Πρώτον, σε επίπεδο ευρωπαϊκού εξαμήνου και δεύτερον, κατά τους συνήθες χρόνους για την προετοιμασία του εθνικού προπολογισμού. Δεν θέλουμε να κλέψουμε καθόλου τίποτα από τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες του ε, εκάστοτε Εθνικού Κοινοβούλου. Αντίθετα, θέλουμε να τους δώσουμε έναν τρόπο ώστε να μπορούν να παρεμβαίνουν πιο αποτελεσματικά στο ευρωπαϊκό σχέδιο. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα να το κάνουμε στο προεξάμεινο και δεύτερον κατά την παραδοσιακή συζήτηση και τον προπολογισμό. Γι' αυτό μιλώ για προπολογισμό, για προπολογισμό σε δύο φάσεις. Ευρωπαϊκή φάση, εθνική φάση. Άρα, αυτό που βλέπετε εδώ, σε αυτό το τόσο σύντομο κείμενο, είναι μια πολύ σύντομη γνωμοδότηση και αφορά στοιχεία από αυτό το δημοκρατικό ελέγχο διαδικασία. Και θεωρώ πως σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι αντικείμενο μια διοργανική ε, συμφωνία, δηλαδή Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο, Συμβουλίο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα τρία θεσμικά όργανα θα πρέπει να καταλήξουν σε μια συμφωνία που να ορίσει τον τρόπο με τον οποίο θα κυλάει το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, ώστε να είναι απόλυτα σαφές και για μας και για τα εθνικά κοινοβούλια ότι συμμετέχουμε σε μια καθοριστική στρατηγική για την έγκριση των εθνικών προπολογισμών. Έπειτα, άλλα ζητήματα που αφορούν τη διάδοση των πληροφοριών ε, για την αύξηση της συμμετοχής του Ευρωπαίου πολίτη στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο την ανάγκη η Κομισιόν να εξηγεί και να δικαιολογεί τους λόγους του οποίους έκανε κάποιες ε, πολιτικές επιλογές και επέλεξε με έναν τρόπο προτεραιότητες και έπρεπε ε, την ευθύνη να εξηγεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που διαφωνεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι αποκλήσεις λοιπόν, οι αφιστάμενες απόψεις που μπορεί να έχουμε θα πρέπει να τεκμηριώνονται πάντοτε. Αυτά είναι τα κύρια σημεία αυτής της γνωμοδότησης. Και πάλι θέλω να πω ότι αφορούν καθαρά θεσμικά ζητήματα και όχι τα θέματα ουσίας για τις πολιτικές και οικονομικές επιλογές, δημοσιονομικές επιλογές. Αυτά είναι θέματα αρμοδιότητας Επιτροπής ΕΚΟΝ. Ευχαριστώ. Ε, ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Ρανζέλο. Ο λόγος τον κύριο Κουρμάη. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Να κάνω κάποια σχόλια γρήγορα. Να ευχαριστήσω για τη δουλειά που έγινε για τη γνωμοδότηση αυτή και την Ελίζα Φρέρα. Να θυμηθούμε ότι στην Ουγγρική Προεδρία Είχαμε αντίστοιχα πολλή δουλειά. Όταν συζητούσαμε το six pack, ε, κάναμε πολλή δουλειά και συνειδητοποιήσαμε ότι έχει πάρα πολλά να κάνει η Ευρώπη αν θέλουμε να επιβιώσουμε αυτή τη κρίση. Για μένα λοιπόν το ευρωπαϊκό εξάμεινο είναι πολύ σημαντική συνιστόσα του όλου πακέτου. Αν θέλουμε να ξεπεράσουμε την κρίση και να αποφύγουμε στο, μάλλον, στο μέλλον να ζήσουμε τα ίδια. Βεβαίως τους τελευταίους μήνες έχουν παρθεί κάποιες αποφάσεις ε, αλλά εγώ πιστεύω ότι ο οικονομικός διάλογος θα πρέπει να συνεχιστεί και θα πρέπει να συνεχιστεί, ε, να συζητηθεί και το θέμα της δημοκρατικής εκπροσώπησης ή του δημοκρατικού ελλείμματος και από εκεί και πέρα θα πρέπει να ε, συνεχίσουμε το διάλογο πριν να, να προπάμε τελικά στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το οποίο θα πρέπει να αποφασίσει αναχώρα ορισμένα πράγματα. Χρειάζεται πολλή δουλειά, χρειάζεται δουλειά με σαφήνεια, με διαφάνεια, διαφορετικά θα, δεν θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις ευθύνε που έχουμε έναντι των πολιτών μας, των κυβερνήσεών μας, των χωρών μας. Και πιστεύουμε ότι θα μπορούσαμε, θα ήταν καλό πριν από το αερινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάθε χρόνο να γίνεται μια διακοινοβουλευτική συνάντηση μεταξύ ημών και των συναδέλφων από τα κράτη-μέλη. Αυτό θα ήταν καλό. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Νταφ. Δεν είμαι βέβαιος ότι χρειάζεται μια τέτοια μεταβατική συμφωνία. Έχουμε μια συμφωνία πλαίσιο για τον τρόπο με τον οποίο συνεργαζόμαστε με τα άλλα θεσμικά όργανα και δεν θα ήθελα η εποπουτία της οικονομικής διακυβέρνησης να καταλήξει τελικά να γίνει πολύ πλοκή και βαραφορτωμένη. Θέλω να το ξανασκεφτώ και να μιλήσω και με συναδέλφους στην Επιτροπή Εικόνων για να δω τι ακριβώς σκέφτονται και εκείνοι έκθεση αυτή θα έπρεπε να εξεταστεί στα πλαίσια της Δημέτρου για να φανεί ότι χρειάζεται απαραίτητος περισσότερη συμμετοχή του Κοινοβουλίου. Ίσως λοιπόν να χρειαστεί κι άλλη συζήτηση για τα περιθώρια ώστε να μπορέσει εκεί ο Πάολο να με πείσει. Γιατί εγώ νομίζω ότι έχουμε παρκές πλαίσιο με τη διαθεσμική συμφωνία. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν ο συνάδελφος ο οποίος Άγγελ θέλει να πει κάτι. Πολύ σύντομα παρακαλώ. Να είμαι πολύ σύντομος. Ε, θέλω απλά να πω ότι ευχαριστώ του συναδέλφους για την προσοχή που επιδεικνύουν και πράγματι θα λάβω υπόψη αυτό που είπε η κυρία Κουρμάη και ο κύριος Ντάφ. Ναι, είναι καλό να, να το δούμε αυτό το θέμα περαιτέρω, να αμφίβολα. Ειλικρινά θέλω να πω ότι θέλησα με αυτή τη γνωμοδότηση να φέρω το θέμα και σε επίπεδο εθνικών κοινοβουλίων. Πολύ συχνά τα κοινοβούλια μιλούν για ευρωεξάμεινο χωρί να γνωρίζουν γιατί πράγμα μιλάμε και χωρί να γνωρίζουν πόσο σημαντικό Μα σημαντικό ρόλο και καθοριστικό ρόλο έχει το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και άρα θα πρέπει τα κοινοβούλια mm. να μπορέσουν να, ε, μπουν στο παιχνίδι νωρίτερα. Αν μπορέσουν να το κάνουν αυτό και να επηρεάσουν τα πράγματα νωρίτερα, σίγουρα η πολιτική τους επιρροή σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα είναι πολύ σημαντικότερη από αυτή που έχουν σήμερα. Και επειδή μίλησα για διοργανική συμφωνία, μίλησα για κάτι τέτοιο για να μπορέσουμε να διευκρινίσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται αυτό και να δημιουργηθεί ο χώρο. Όχι μόνο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και για τα Εθνικά Κοινοβούλια να έχουν ρόλο εν προκειμένου. Ναι, ίσως χρειάζεται να γίνει αυτό με έναν καλύτερο τρόπο και καλό είναι να συνεχιστεί αυτή η συζήτηση και φυσικά λαμβάνω υπόψη ναι, δεόντως ε, και την παρατήρηση του κυρίου Ντάφ. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ λοιπόν. Από εδώ και πέρα τι γίνεται για αυτή τη νομοδότηση, επειδή το χρονοδιάγραμμά μας μας πιέσει και προκύπτουμε γρήγορα, θα πρέπει κατά εξαίρεση ψηφοφορία να γίνει στις 21 Ιανουαρίου και άρα να ορίσουμε και την κατευθυντική ημερομηνία για τις ε, τροπολογίες στις 8 ε, Ιανουαρίου, 12 το μεσημέρι. Και επειδή είναι δύσκολη αυτή η περίοδος λόγω Χριστουγέννων να τα πούμε ε, είτε εδώ είτε στο Σασβούργο, για πρώτη φορά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ηλεκτρονική υπογραφή για την υποβολή αυτών των τροπολογιών. Συμφωνείτε λοιπόν, ψηφοφορία στις 21, 21 Ιανουαρίου, ψηφοφορία λοιπόν στις 5 το απόγευμα πριν τους συντονιστές και τροπολογίες έως 8 Ιανουαρίου και, και ηλεκτρονικά μπορείτε. Αν συμφωνείτε, να περάσουμε τώρα στην εδρία των συντονιστών. Merry Christmas. Joyeux Noël. Joyeux Noël.